Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η οδηγία που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντάσσεται στο πλαίσιο ορισμένων εγγράφων στα οποία είχαμε ήδη την ευκαιρία να εμβαθύνουμε σε άλλες ευκαιρίες, το CARS 2020 για παράδειγμα, που έχει ως στόχο την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και την αηφορία των επενδύσεων σε καθαρές προηγμένες τεχνολογίες καθώς και στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Κομισιόν του 2010 υπέρ της υποστήριξης των πράσινων οχημάτων για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Επίσης, σε αυτή την ανακοίνωση τονίζονται οι ελλείψεις ε, του κοινοτικού πλαισίου, κυρίως για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και για την υποστήριξη της προώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος αυτής της νέας οδηγίας, αυτό που επιθυμεί η Κομισιόν, είναι η υλοποίηση μια ελάχιστης ε, υποδομής για τα εναλλακτικά καύσιμα και η εφαρμογή τεχνικών προτύπων κοινών σε κοινωτικό επίπεδο. Η διατήρηση της ευρωπαϊκής επιρροχής στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη ε, και στα πλοία, διότι αφορά επίσης και τα καύσιμα για τα πλοία. Να μειωθεί η εξάρτηση όσον αφορά το πετρέλαιο για τις μεταφορές και μείωση των αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2050. Αυτή η πρόταση οδηγίας καθορίζει προδιαγραφές ε, για εθνικά στρατηγικά πλαίσια. Δεσμεύει τα κράτη-μέλη να ορίζουν ε, δεσμεύσεις ε, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες για την ανάπτυξη καυσίμων για τις μεταφορές. Προβλέπει επίσης ε, υποδομές για εναλλακτικά καύσιμα και υλοποίηση συγκεκριμένων κοινών τεχνικών για τις εν υποδομές. Επίσης καθιστά υποχρεωτική την ελάχιστη κάλυψη με υποδομές για τον ανεφοδιασμό με ηλεκτρισμό, υδρογόνο και φυσικό αέριο. Δεν πρέπει λοιπόν να κάνουμε το λάθος να θεωρούμε ότι αυτό το κείμενο αναφέρεται μόνο στα ηλεκτρικά οχήματα αναφέρεται και σε όλα τα εναλλακτικά καύσιμα φυσικό αέριο, υδρογόνο και ηλεκτρισμό. Επίση, προτείνει να ορίζεται ο ελάχιστο αριθμό σημείων αναφοδιασμού ανακρατός μέλο βάσει εθνικών στόχων όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα. Στο κείμενο τη οδηγία προβλέπεται ότι το 10% αυτών των σημείων εφοδιασμού θα πρέπει να είναι προσπελάσιμο σε όλου, τουλάχιστον το 10%. Επίση, προβλέπει μια σειρά προδιαγραφών όσον αφορά την ελάχιστη απόσταση μεταξύ σημείων ανεφοδιασμού ανάλογα με τους διάφορους τύπους εναλλακτικών καυσίμων, υδρογόνο, φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο και πεπιεσμένο φυσικό αέριο. Είτε δηλαδή για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για τα οχήματα κίνησης, όσο και για την αυσιπλοεία. όπως και για το φυσικό αέριο για τις οδικές μεταφορές. Ένα κομμάτι αυτού του κειμένου αφορά την ενημέρωση προς τους καταναλωτές. Το πώς οι πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές θα είναι πιο σαφείς, πιο απλές όσον αφορά τη συμβατότητα μεταξύ καυσίμων και οχημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά στους σταθμούς αναφοράς, ε, στα εγχειρίδια των οχημάτων και στα ίδια τα οχήματα. Ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να συζητηθεί αφορά τις κατεξοδότηση πράξεις Όπου έχει γίνει αρκετή συζήτηση στην Επιτροπή μα, εκεί θα προβλέπεται η δυνατότητα η Κομισιόν να επανεξετάζει την γκάμα εναλλακτικών καυσίμων, την κάλυψη των υποδομών και την υλοποίηση των συγκεκριμένων τεχνικών για τα καύσιμα και τις αντίστοιχες υποδομές. Στη φάση ακρόασης που διεξάγω εγώ αυτή τη στιγμή ως εισηγητής, ε, αντιλήφθηκα μέχρι στιγμής ότι έχουμε μια καλή ε, αφετηρία, ένα καλό εφαλτήριο βάσει της πρότασης της Κομισιόν. Φυσικά υπάρχουν προσδοκίες από τους φορείς του τομέα. Θα πρέπει με αυτή την οδηγία να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση που θα ικανοποιεί πολλούς τομείς, διότι εδώ εμπλέκονται όχι μόνο οι παροχής ενέργειας, όχι μόνο οι βιομηχανίες ε, που κατασκευάζουν οχήματα γενικότερα. Εμπλέκονται επίσης τα κράτη-μέλη κατά τρόπο ουσιαστικό επειδή από αυτά εξαρτάται ο ορισμός του πλήθους των στόχων των στρατηγικών πλαισίων. Εμπλέκονται επίσης η παραγωγή των ίδιων των υποδομών όπως τα ηλεκτρικά κολονάκια. Πολλοί λοιπόν τομείς ε, εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και έτσι εμείς πρέπει να διεξαγούμε σε βάθος ακρόαση ώστε οι στόχοι που προβλέπει αυτό το κείμενο να συμπερφώνονται με τις προσδοκίες της αγοράς και να είναι παρκώς φιλόδοξοι σε σχέση με τους στόχους που έχουμε θέσει πολλάκες. Δεν πρέπει λοιπόν να επικεντρώθουμε μόνο στα ηλεκτρικά οχήματα, αλλά να λάβουμε υπόψη και τις υπόλοιπες πτυχές των υπόλοιπων καυσίμων που εξετάζονται σε αυτό το κείμενο. Υπάρχει μια πτυχή που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και να αξιολογήσουμε σίγουρα με την Λιθωνική Προεδρία διότι αυτή θα ολοκληρώσει αυτό το κείμενο καθώς αυτός ο φάκελος δεν θα μπορέσει δεν θα προλάβει να το τελειώσει η Ιρλανδική Προεδρία θα πρέπει να δούμε τη συμβατότητα των στόχων με την πραγματικότητα που ισχύει στα διάφορα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν οι προθεσμίε υλοποίηση τη οδηγία θα αποτελούν σημαντικό κομμάτι τη συζήτηση που πρόκειται να έχουμε. Τίθεται επίση το ζήτημα των παραρτημάτων, διότι στα παραρτήματα περιλαμβάνεται μια σειρά δεδομένων, συγκεκριμένων τεχνικών, τεχνικών προδιαγραφών, σημαντικών για διάφορους τομείς και διάφορες βιομηχανίες που αφορά αφορούν αυτές οι διατάξεις. Ε, τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται αυτή τη στιγμή για τη συζήτηση αυτής της οδηγίας προβλέπουν ε, παράδοση του σχεδίου έκθεσης τον Ιούλιο, ανάλυση της έκθεσης το Σεπτέμβριο και ψηφοφορία στην Επιτροπή στα μέσα Νοεμβρίου. Μετά από μια πρώτη φάση ακρόασης ε, και πιστεύω οι συντονιστέ θα μα δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε μια μήνυα ακρόαση ε, εντός τη Επιτροπής. Πιστεύω τότε θα μπορέσουμε να μπούμε στην ουσία τη συζήτηση και να ε, έχουμε μια αποτελεσματική, ε, να κάνουμε μια αποτελεσματική δουλειά. Ευχαριστούμε κύριε Φιντάντσα, ο κύριος Αλχαντροή. Dank u voorzitter. Ehm, ik wil om te beginnen συνάδελφος έπρεπε να είχε πάει στην Λιθουανία για να προετοιμάσει την Λιθουανική Προεδρία και ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι παρούσα στη συζήτηση διότι πραγματικά θεωρεί πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Ενδιαφερόταν εδώ και πολλά χρόνια για το θέμα των εναλλακτικών καυσίμων και για τις θαλάσσιες μεταφορές και για τις ποτάμιες μεταφορές. Η χρήση του GNL επιτρέπει να μειωθούν οι εκπομπές οξυδίου του αζότου, την, ενώ εκμηδενίζει τις εκπομπές θείου. Πρόκειται για ένα σημαντικό ε, θετικό στοιχείο σε περιοχές όπως η Βαλτική και η Βόρεια Θάλασσα, που είχαμε μεγάλες εκπομπές πέρσι. Μέχρι τώρα οι εφοπλιστές μας έλεγαν ότι η τεχνολογία GNL δεν είναι επιλογή, ενώ όσο δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα βρίσκουν GNL στα λιμάνια στα οποία φτάνουν. Άρα δεν υπήρχε ενδιαφέρον να υπάρξει υποδομή GNL παρά μόνο όταν χρειάζονται τα σκάφη. Η πρόταση της Επιτροπής είναι καλή λύση για να βγούμε από την, ε, ε, ε, από την, από την διαδικασία αυτή. Αυτό θα επιτρέπει την χρησιμοποίηση της τεχνολογίας αυτής με επιθετικό τρόπο. Επίσης εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για το πρόγραμμα δράση που δημιουργήσε η Επιτροπή για, με την ε, οδηγία για τα, εναλλακτικά καύσιμα και ε, θεωρεί θετική την έκθεση Φιντάντς. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Lichtenberger for the Greens. είναι πολύ φιλόδοξη. Περιλαμβάνει μια σειρά στόχων, εξαιρετικών στόχων, μείωση των εκπομπών από τις διάφορες, ε, τα διάφορα είναι στόχος που συμμεριζόμαστε όλοι. Όταν βλέπω την μείωση της περιεκτικότητας θείου για τις θαλάσσιες μεταφορές για παράδειγμα, θα έλεγα ότι πρόκειται για εξαιρετικό στόχο. Το πρόβλημα ωστόσο Πρόεδρε, έγκυται στο, να δούμε κατά πόσον θα δώσουν αποτέλεσμα οι προθέσεις αυτές. Και εγώ έχω ορισμένε επιφυλάξεις που θα τις αναφέρω. Όλο το χρηματοοικονομικό στοιχείο, για παράδειγμα. Έχουμε κάποιους πίνακες στο παράτημα, αλλά δεν με πείθουν. Δεν με πείθουν ότι είναι στέρεα οικονομικά αυτά το προπολογισμό των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών εξαρτάται για παράδειγμα από τη συνολική συζήτηση για τι δημοσιονομικέ προοπτικές τη Ένωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πρώτο λοιπόν πρόβλημα η χρηματοδότηση και δεν μιλώ μόνο για, τη, το κονδύ, για τα κονδύλια της Ένωσης αλλά και την οικονομική συμβολή των κρατών μελών και την πολιτική τους βούληση διότι ωραίο είναι να κάνουμε προτάσεις φιλόδοξες αλλά χωρίς την συνεργασία των κρατών μελών δεν θα πετύχουμε τίποτα. Θα ήθελα λοιπόν να έχω κάποιες διευκρινήσεις από την Επιτροπή για το σημείο αυτό. Την χρηματοδότηση και ιδίω τη συμβολή, τη συνεισφορά των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Δεύτερο σημείο προβληματικό για μένα είναι η πρίζα του ρεύματος του αυτοκινήτου. Μας παροτρύνουν προς μια γερμανική λύση ευρωπαϊκά δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι η καλύτερη λύση. Υπάρχει το Ιαπωνέζικο μοντέλο που λειτουργεί με τελείως διαφορετικό τρόπο. Πώς θα δουλέψουμε. Φαντάζομαι ότι σε ό,τι αφορά την πρίζα του ρεύματο θα υπάρχουν κάποια σημεία επαναφόρτησης που όπως και στις αντιλίες βενζίνης μπορεί να βάλεις δίζελ ή βενζίνη, τέλο πάντων θα έχει ένα αντίστοιχο. Μια μπρίζα γερμανικού χαρακτήρα ή μια μπρίζα γιαπωνέζικου χαρακτήρα. Είναι μια συζήτηση πολύ σημαντική, Πρόεδρε, που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ή να αποφασίσουμε έτσι ε, χωρίς πολλή συζήτηση. Και τρίτον, τι θα κάνει το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εξηγώ τι θέλω να πω. Όταν πηγαίνω στο Στρασβούργο με αυτοκίνητο, αν πάρω ένα καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα μπορώ να φορτίσω το αυτοκίνητό μου στο πάρκινγκ του Στρασβούργου ή των Βρυξελών. Αν μη τι άλλο θα έπρεπε να καθαρίσουμε πρώτα τις δικές μας ε, ευθύνες. Θα αλλάξει το Κοινοβούλιο την υποδομή του. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο θα ξεκινήσουν δίνοντας το καλό παράδειγμα, αλλάζοντας τις υποδομές τους για, τις εναλλακτικές, ε, για τα εναλλακτικά καύσιμα. Και κλείνω. Ωραία πρόταση, μακρύς ο δρόμος και γεμάτος εμπόδια. Ελπίζω σήμερα ή αργότερα η Επιτροπή να μας διευκρινίσει μια σειρά προβληματικών ερωτηματικών στοιχείων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρίκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για αυτή την πρόταση συνάδει με τις προτεραιότητες της ομάδας μας δεν ακούω αγγλικά μέσω του αγγλικού καναλιού λέει ο πρόεδρος Dominic, μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι εντάσσεται αυτή η οδηγία σε ένα γενικό πλώσιο. Υπάρχουν δύο διαφορετικά προβλήματα. Το ένα ανέφεραν δύο προηγούμενοι ομιλητές είναι το οικονομικό πρόβλημα. Ήθελα να υπενθυμίσω ότι στο μηχανισμό συνδέοντα την Ευρώπη έχει προβλεφθεί στι οριζόντιε προτεραιότητε. Φυσικά υπάρχουν αβεβαιότητε όσον αφορά τη χρηματοδότηση των διαθέσιμων όγκων ε, των διαθέσιμων ποσών, τα ποσοστά, αλλά σίγουρα οι πόροι δεν επαρκούν, οι πόροι δεν επαρκούν στο Connecting Europe. Και υπάρχει κάτι που μας ενοχλεί. Εάν σε αυτό το μηχανισμό Connecting Europe έχουμε το χρηματοδοτικό μέσο και ξέρουμε ότι αυτό δεν φτάνει, δημιουργείται ένα πρόβλημα. Αυτή η χρηματοδότηση μέσω του Connecting Europe θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας. Το δεύτερο που μου φαίνεται εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτή η οδηγία εντάσσεται στο γενικότερο ενεργειακό μείγμα. Διότι μιλάμε για εναλλακτικέ μορφές ενέργειας, για οτιδήποτε κινείται και οτιδήποτε πετάει και οτιδήποτε πλέει, αλλά όλο αυτό εντάσσεται σε μια γενική ενεργειακή κατανάλωση. Πρώτο παράδειγμα όσον αφορά το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εάν για παράδειγμα το σύνολο του γαλλικού στόλου περάσει σε ηλεκτρικά οχήματα, χρειάζονται καμιά εικοσαριά ε, πυρηνική σταθμή ενέργειας για να μπορέσουν να τροφοδοτηθούν. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η γενική προμήθεια στο πλαίσιο του ενεργειακού μείγματος και το θέμα των πόρων. Αυτό θα επηρεάσει το γενικό σχέδιο, δηλαδή τι ποσότητες ενέργειας χρειαζόμαστε και τι τρόπους ανεφοδιασμού. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι επίσης η αποθήκευση της ενέργειας. Όταν μιλάμε για ανεφοδιασμό με υδρογόνο, εγώ αντιλαμβάνομαι δίκτυα υδρογόνου, το οποίο δεν μου φαίνεται εφικτά για διάφορους λόγους, οικονομικούς, υποδομών. Ε, πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι σταθμοί υδρογόνου ε, μπορούν να αποτελέσουν λύση και για την αποθήκευση ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό το θέμα δεν μπορούμε να μην το συζητήσουμε στο πλαίσιο αυτή τη οδηγία. Συνεπώ πρέπει να ορίσουμε τη θέση μα όσον αφορά το χρηματοδοτικό κομμάτι και το κομμάτι του ενεργειακού μείγματο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εναλλακτικέ μορφέ ενέργεια χωρί να ξέρουμε από πού θα τι πάρουμε, πώς, με ποιο τρόπο θα τι μεταφέρουμε και πώ θα τι κατανείμουμε. Μια άλλη παρατήρηση, όπως ανέφερε ο Βαντάλεν για την τυποποιημένη πρίζα, βλέπουμε γίνονται συζητήσεις για τις τυποποιημένες ε, πρίζες ε, ε, του τύπου 2 και άλλες χώρες θέλουν τον τύπο 3 που περιλαμβάνει μια επιπλέον ασφάλεια και δεδομένου του επιχείρηματος ασφάλειας φαίνεται να είναι ισχυρό το επιχείρημα. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε μια πρόταση σε αυτή την οδηγία επί του θέματος για να δούμε τελικά θα έχουμε δύο-τρεις ε, πρίζες τυποποιημένες σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το ρυθμισμένο πλαίσιο. Δεν πρέπει να το αφήσουμε σε κρεμότητα. Κάτι άλλο που θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού που υπάρχουν ήδη. Μπορεί να καταλήξουμε σε ένα παράδοξο όπου οι άνθρωποι που ήταν πρωτοπόροι σε αυτό το θέμα να υποστούν κυρώσεις. Ουσιαστικά οι νέες ρυθμίσεις που θα να τους επιβάλλουν τιμωρίες θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε μεταβατικά μέτρα για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Αυτέ ήταν οι παρατηρήσει που ήθελα να κάνω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Λίχτεμπεργκερ. Ja, herzlichen Dank. θέλω να επαναλάβω κάποιες από τις παρατηρήσεις ε, του σκιώδου του κ. Βαντάλεν και να κάνω και κάποια σχόλια. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να δούμε μείωση των εκπομπών παντού. Το πρόβλημα με την έκθεση της Επιτροπής, ωστόσο, είναι πραγματικό ότι έχω μείνει αποσβολωμένη. Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που δεν έλαβε υπόψη. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις και πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις. Πηγαίνετε στην πλατεία εδώ του Λουξεμβούργου. Θα δείτε δίπλα στην τράπεζα ING υπάρχουν δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν, δεν έχουν κινηθεί ποτέ. Προφανώ δεν έχουν δεν λειτουργεί μπαταρίε. Τι πρακτική επίπτωση έχουν όλα αυτά. Μιλάμε για τεράστιε επενδύσει, Ήδη αναφέρθηκε το οικονομικό κομμάτι. Πραγματικά μα ανησυχούν μια σειρά δηλώσεων. Η Επιτροπή εξειδικεύει τέσσερα, τέσσερις κατηγορίες ε, ισχύω των αυτοκινήτων. Ποια είναι όμως, γιατί τέσσερα, είναι τα σωστά τέσσερα ή σωστές τέσσερις ε, κατηγορίες ανάλογα με το κλίμα ή τη γεωγραφική κατάσταση μιας χώρας. Τι γίνεται με την ενέργεια που παράγεται από τα, από τα πυρηνικά απόβλητα. Βάζει ένα στόχο, 2020. Τώρα είμαστε το 2013. Δηλαδή, σε κάποιες χώρες δεν μπορούν να προχωρήσουν. Προφανώς μπορούν να προχωρήσουν. Αλλά για μένα το όλο θέμα είναι πώς θα εξελιχθούμε. Πώς θα εξελιχθούμε με την εξέλιξη τη τεχνολογία. Δεν είναι θέμα οδηγία ή κανονισμού. Γιατί πιστεύω ότι αυτό που δεν θέλουμε είναι να έρθει η Επιτροπή και να αποφασίσει τι θα είναι στάνταρ και τι δεν θα είναι. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι τι θα κάνει η αγορά. Ήδη μιλήσαμε για το ότι δώσαμε τελικά, βάλαμε σε μειονεκτικότερη θέση αυτούς που ξεκίνησαν, ε, ε που ξεκίνησαν νωρίς. Ε, μιλάτε για 144 χιλιόμετρα ε, αντλίες. Πού έχετε πάει στη Σκωτία να δείτε ότι υπάρχουν αποστάσεις πολύ μεγαλύτερες. Τι θα γίνει, θα βάλουμε αντλίες εκεί που δεν υπάρχει τίποτα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να καθορίζουν τη δική τους πολιτική ανάλογα με τις ανάγκες τους, πρακτικά και κάνουν δουλειά, το ψάχνουν αυτό, είναι ένα κοινό ζήτημα, αλλά πρέπει να σεβαστούμε την επικουρικότητα, την γεωγραφική κατάσταση, να είμαστε ευέλικτοι και να έχουμε μείωση των εκπομπών με κόστο αποτελεσματικό τρόπο. Θα έπρεπε η Επιτροπή να το ξαναδεί, να ξαναδεί τις, τις αποστάσεις, να ξαναδεί τις ημερομηνίε και να απαντήσει στα ερωτήματα που τέθηκαν για τη χρηματοδότηση και τις το πόσο πρακτικό είναι αυτό που προτείνει. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά πρόημο και θα καταπέσει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπράτμπορν. Ήδη αυτά που θέλατε να πείτε έχουν υποθεί. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο κ. Βαντάλλαν και η κυρία Φώστερ και ο κ. Ρικέη. Υπάρχουν κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την κυρία Φώστερ και θα ήθελα να το τραβήξω και λίγο παραπέρα. Πιστεύω ότι είναι από τις πιο λανθασμένα σχεδιασμένες προτάσεις που έχουμε δει εδώ και πολύ καιρό από την Κομισιόν. Και πάλι εδώ έχουμε έναν από τους τομείς όπου προσπαθούμε να προκαταβάλουμε μία λύση για ένα πρόβλημα το οποίο ειλικρινά δεν υπάρχει ακόμα. Όπως γνωρίζετε, αφενός η τεχνολογία έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της. Βρίσκεται υπό εξέλιξη. Δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξει αυτό το είδος τεχνολογίας. Ε, η κυρία Λέχτεμπεργκ ε, ανέφερε όλα τα ζητήματα αυτά που ανέφερε και εγώ συμφωνώ μαζί της παραδόξως. Δεν πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις σε ανθρώπους πρωτοπόρους στην αγορά. Ωστόσο, αυτό που εδώ που βλέπουμε μπροστά μας προδιαγράφει ακριβώς αυτό. Είναι απαράδεκτο κατά τη δική μου άποψη. Αυτή η προσέγγιση που προσαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις δεν πρόκειται να λειτουργήσει διότι σε κάθε κράτος μέλος θα εκφραστούν διαφορετικές απόψεις και θα υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές όσον αφορά το ενεργειακό μείγμα για τις διάφορες μορφές μεταφορών. Και αυτό εντάσσεται στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Δεν μπορεί να το ορίσει Κομισιόν. Δεύτερον, μιλώντας, ε, ανέφεραν διάφοροι ε, ελάχιστα ε, πλήθη σταθμών φόρτωσης, φόρτισης κατά μήκος του δικτύου. Πολλοί θα πούν ότι εγώ είμαι τόσο γέρος που θυμάμαι τα πρώτα αυτοκίνητα, αλλά ειλικρινά δεν θυμάμαι. Αλλά όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα αυτοκίνητα και χρειαζόταν βενζίνη, οι άνθρωποι έλεγαν ότι χρειάζεται ένα βενζινάδικο κάθε δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα. Αλλά αυτό το άφησαν τελικά στην αγορά. Και εκεί όπου υπήρχε ζήτηση, η αγορά ήρθε να καλύψει αυτή τη ζήτηση. Το να αρχίσουμε τώρα να θέτουμε αυτές τις ελάχιστες απαιτήσει είναι αστείο κυρίως εφόσον είμαστε αβέβαιοι για το ενεργειακό μείγμα του κάθε κράτους μέλους στην Ευρώπη. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω και υπάρχει αυτό στο σχέδιο πρότασης και μάλιστα θέλω να θέσω μια ερώτηση εδώ στην Κομισιόν ή στον εισηγητή. Αναφέρεται στο γεγονός ότι όλο αυτό θα χρηματοδοτηθεί μερικώς από το πρόγραμμα των διευρωπαϊκών δικτύου. ή από το Connecting Europe, από το Μηχανισμό Σύνδεοντα στην Ευρώπη, που ίσω να είναι καταλληλότερο μέσο, κατά την άποψή μου, για μερική χρηματοδότηση. Πώ θα γίνει όμω αυτό, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και συνεπώ δεν γνωρίζουμε τι χρήματα θα υπάρχουν στον Κορβάνα. Το να προτείνουμε λοιπόν νέε εναλλακτικέ μεθόδου χρηματοδότηση όταν δεν γνωρίζουμε με σιγουριά τις λεπτομέρειες αυτού του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου, για μένα είναι εντελώς ε, ε, παρανοϊκό. Πρέπει να... Δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα καταλήξουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Πρέπει να περιμένουμε την κατάληξή τους, την έκβασή τους, να δούμε τι συνέπειες θα έχει αυτό για το πρόγραμμα διευρωπαϊκών δικτύων και συνδέοντας την Ευρώπη και τότε θα μπορέσουμε να κρίνουμε λογικά κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμμετέχει στην επίλυση αυτών των ζητημάτων. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σημείο κλειδί το οποίο χρειάζεται να επιληθεί πριν προχωρήσουμε περαιτέρω όταν μιλάμε για τέτοια ζητήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φιντάντσα. Ξέρω ότι θέλετε να απαντήσετε. Θέλετε να απαντήσετε τώρα ή να αφήσουμε πρώτα την Κομισιόν. Περιμένω, με περιμένουν στην Επιτροπή για μια σημαντική συνάντηση από την οποία δεν μπορώ να φύγω. Κατέγραψα τις παρεμβάσεις όλων σας ε, περιμένω να συναντήσω το συντομότερο δυνατό τους και συγκητές για να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση εν ώψη και να έχουμε ένα σχέδιο κειμένου. Συγγνώμη που φεύγω τρέχοντας. Η Επιτροπή θέλει το λόγο. επαναλάβω μάλλον αυτά που είπε ο εισηγητή ότι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Μήνυ ακρόαση 18 Ιουνίου. Εάν το εγκρίνει αργότερα η συνάντηση των συντονιστών, αυτή είναι η πρόταση πάντω. Παρουσίαση του σχεδίου έκθεση στις 16-17 Σεπτεμβρίου, προθεσμία τροπολογιών 1η Οκτωβρίου και εξέταση των τροπολογιών 4-5 Νοεμβρίου με ψηφοφορία στην Επιτροπή 14 Νοεμβρίου. Μπορεί λοιπόν να φαίνεται ότι έχουμε ακόμα πολύ καιρό μπροστά μας. Είναι σημαντικό να έχουμε τις προθεσμίες υπόψη μας. Ευχαριστώ. Επόμενο θέμα. Παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης για τα καύσιμα και την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές έμεση αλλαγής της χρήσης γης. Ε, γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η υπεύθυνη είναι η κυρία Βουέλ. Παρακαλώ. Σαμπίν Βίλς. Ευχαριστούμε πολύ για το ΕΛΚ, ο κύριος Μπορισόφ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η προώθηση των βιοκαυσίμων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την ενεργειακή και κλιματική στρατηγική και αποτελεί εργαλείο μέτρησης της πρόοδου του περιβαλλοντικού τομέα. Αφορά μεγάλο ποσοστό Τη της μείωσης εκπομπών. Ταυτόχρονα η χρήση των βιοκαυσίμων έχει δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης στην Ευρώπη και βοηθάει τις χώρες στην πρόθεση των τεχνολογικών εξελίξεων. Ωστόσο, τα βιοκαύσιμα έχουν και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις. Η Κομισιόν κάνει μια νομοθετική πρόταση για την ελαχιστοποίησή τους, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα πόσο σημαντικό είναι η ενθάρρυνση ε, χρήση των ε, βιοκαυσίμων. Θα μπορούσα να συζητήσω, κυρία Μπορισόφ, να μιλάτε και πιο αργά, ώστε να μπορούν οι διερμηνείς. Τα βιοκαύσιμα έχουν και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις. Η Κομισιόν έκανε μια νομοθετική πρόταση για την ελαχιστοποίησή τους. Αναγνωρίζω, ενώ αναγνωρίζετε πόσο σπουδαίο είναι να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση προηγμένων βιοκαυσίμων που έχουν σχεδόν μηδενικές ε, εκπομπές αερίων θερμοκηπίων και σε σχέση αυτό με την αλλαγή χρήσης γης είναι σημαντικό να μην ε, δημιουργήσουμε κυρώσεις για το τρέχον σύστημα. Η Προστατεύοντα τι υπάρχουσε επενδύσει και στέλνοντα ένα μήνυμα στην αγορά ότι η εξέλιξη θα πρέπει να βασιστεί στα προηγμένα βιοκαύσιμα. Αυτό είναι κατά την άποψή μου εξαιρετικά σημαντικό δεδομένη τη σημερινή οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Η παραγωγική δυνατότητα προηγμένων βιοκαυσίμων στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι πολύ περιορισμένη και η απαραίτητη επένδυση που απαιτείται για την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον η πολιτική της Ευρώπης δημιουργήσει ένα σταθερό και παραγωγικό ε, ρυθμιστικό πλαίσιο που θα παρέχει βεβαιότητες στους επενδυτές. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι η χρήση των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι πολύ καλή ιδέα και πρέπει να ληφθούν οι υπόψη και οι επενδύσει που πρέπει να γίνουν σε ορισμένε χώρε τη πρώην Ανατολική Ευρώπη, διότι εκεί οι επενδύσει πρέπει να είναι πολύ μεγάλε και οι σημερινέ οικονομικέ συνθήκε δεν το επιτρέπουν. Πρέπει να δούμε λοιπόν πόσο εφικτό είναι το 5% ε, κάλυψης της ηλεκτρική ενέργεια στι ιδρυνομικές μεταφορέ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλκαντράουι. Έρχεται ο κύριος Πανιόν. Θα άφησε δύο λεπτά, οπότε αν θέλετε να συνεχίσετε με τους υπόμενους. Ωραία. Κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ. Καταρχάς, συμφωνούμε ότι πρέπει να τηρήσουμε τον στόχο της διατήρησης 10% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και μείωση κατά 6% των εκπομπών ε, αερίου του, αερίου του θερμοκηπίου μέχρι το 2020. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική στόχη πάνω στους οποίους πρέπει να δουλέψουμε. Προς την κατεύθυνση αυτή συμφωνούμε ως προς τους γενικού στόχους που έχει η πρωτοβούλια αυτή. Να περιοριστεί δηλαδή ο, η χρήση των παραδοσιακών βιοκαυσίμων και η βελτίωση των τρόπων παραγωγής, η μεγαλύτερη εγκατάσταση των ε, προηγμένων βιοκαυσίμων που αποκτούν μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με τα παραδοσιακά καύσιμα και εν τέλει η ενίσχυση και ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των κοινοποιήσεων. Επίσης θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να έχουμε κοινοποιήσεις από τα κράτη-μέλη και τους παρόχους που θα ανακοινώνουν ποιες είναι οι εκπομπές των βιοκαυσίμων και τι επιπτώσεις έχουν στην αλλαγή της χρήσης γης. Γι' αυτό πρέπει να είναι συμβατή η ανακοίνωση με την βελτίωση των επιστημονικών δεδομένων που, όπου πρέπει να προχωρήσουμε σημαντικά ακόμα. Επίσης θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να προστατευτούν οι επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει μέχρι τώρα γιατί οι επενδύσεις όλων των επιχειρηματιών έγιναν με την βεβαιότητα και την εμπιστοσύνη ότι οι αποφάσει που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε κάθε κράτο μέλο θα συνεχίζουν να υφίστανται. Κάποιε από τι τροπολογίες λοιπόν τη εισηγήτρια νομίζω ότι πάνε λίγο παραπέρα από αυτό που θέλουμε και από αυτό με το οποίο συμφωνούμε. Ίσως οι τροπολογίες μας θα στραφούν προς αυτά που σας είπα. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει επαρκής εξασφάλιση των κριτηρίων που ανέφερα από την έκθεση και θα δουλέψουμε για να διατηρήσουμε την στάση και θέση που έχει παρουσιάσει η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κύριε Πανιόλ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη χαρά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγήτρια την κυρία Βίλς για την έκθεση της αυτή. Εμείς υποστηρίζουμε απόλυτα τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, λαμβάνοντας υπόψη και τον παραγόντα μείωσης ε, των, ε, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε μια τέτοια οδό όμως όταν έχουμε πολλά αποδεικτικά στοιχεία για τους κινδύνους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτρέψει τη γενικευμένη χρήση των βιοκαυσίμων που ρηπαίνουν περισσότερο από τα κλασικά ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα βιοκαύσιμα δημιουργούν στρεβλώσεις ε, στην αγορά τροφίμων και ειδικότερα οδηγούν σε αύξηση τιμών ορισμένων πρωτονυλών. Η πρόσβαση στα τρόφιμα στις φτωχότερες περιοχές του πλανήτη γίνεται πιο δύσκολη το ίδιο και η διατροφή των ζώων. Όλα αυτά έχουν επιπτώσει στην αλυσίδα παραγωγής. Πιστεύω ότι για λόγους ε, συνοχής ε, το να περιορίσουμε τη συμβολή των βιοκαυσίμων στο 5% από το 10% πιστεύω δεν είναι σωστό παρότι πρόκειται για έναν από τους πυλώνες αυτής της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης η ηλεκτροκίνηση όλων των συστημάτων μεταφορών μας μου φαίνεται ότι δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους που θέλουμε. Χρειάζεται λοιπόν ε, ο ορισμός ανώτατων τιμών ώστε να περιοριστεί η αλλαγή χρήσεων γης. Αλλά δεν πρέπει να ε, αποκλείσουμε άλλα βιοκαύσιμα που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον. Τέλος, ο τρόπος πολλαπλής μέτρησης των βιοκαυσίμων μου φαίνεται ότι ε, είναι, είναι πολύ σωστός, αλλά θα πρέπει να έχουμε έχει έγκυα ώστε να μην στρεβλωθεί αυτό το σύστημα εναρμόνιση στην Ευρώπη τη αντιμετώπιση των περιπτώσεων απάτης, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη ε, στην νομοθεσία και στη σταθερότητα του συστήματος. Αυτά κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τα στοιχεία που ήθελα να παρουσιάσω στα μέλη της Επιτροπής μα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Προφανώς η βασική δουλειά γίνεται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και για να το καταλάβει κάποιος ίσως να χρειάζεται ολόκληρο διδακτορικό. Τι είναι όμως κατά βάση. Κάτι που με ανησυχεί ιδίως. Έχουμε μια σειρά στόχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι θα κάνει το 2020, μέχρι το 2020 ο καθένα μας. Και ένα από τα βασικά θέματα που τίθενται είναι η χρήση γης. Όσο φτάνουμε στόχους και μετά έχουμε χώρες του τρίτου κόσμου που εμπλέκονται σε όλα αυτά, αν εμείς φτάσουμε τους στόχους μας ωραία, δεν είναι σωστό αυτό. Θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση πολύ πιο ρεαλιστική. Δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να τηρούμε τους στόχους των ε, χωρών, δαπανηρούς στόχους για χώρες οι οποίες θα δαπανίσουν πάρα πολύ γι' αυτό ενώ άλλοι δεν θα κάνουν τίποτα. Πιστεύω ότι η οδηγία είναι πολύ περιοριστική, θα αυξήσει το κόστος της συμμόρφωσης και ίσως θα έπρεπε να περάσει ένα μήνυμα για το τι κάνουμε εδώ, διότι έχω την εντύπωση ότι κάποιοι στέκονται εκεί λένε στόχος, στόχος, στόχος, πρέπει να πετύχουμε το στόχο και βεβαίω να πετύχουμε τους στόχους, αλλά νομίζω ότι συνολικά παραγνωρίζουμε την πραγματικότητα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στο τι μπορούμε να πετύχουμε. Εγώ υποστηρίζω την ανάγκη να εξετάσουμε εναλλακτικά βιοκαύσιμα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να το δούμε με πιο ρεαλιστικό τρόπο, όχι εις βάρος χωρών που δεν είναι μέλη της Ένωσης και νομίζω ότι αυτό γίνεται όταν υιοθετήσαμε αυτά, αυτές τις προθεσμίες. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας. Είμαστε κατά κάποιον από τις τοπολογίες 1, 4, 6 που μιλά για συγκομιδές ε, βρόσιμων προϊόντων. Νομίζω ότι αυτό επαναλαμβάνω ότι οι βασικές επιτροπές που θα συζητήσουν το θέμα αυτό είναι περιβάλλοντος και ήτρε, αλλά και εμείς θα πρέπει να το δούμε. Για την Επιτροπή, ο Πίλζεκ από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι ότι οι συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μοιάζουν πολύ με τις συζητήσεις που κάναμε στην Κομισιόν κατά την προετοιμασία της πρότασης. Κατά βάση το πρόβλημα είναι το να λαμβάνουμε υπόψη νέα αποδεικτικά στοιχεία ή πιο σταθερά αποδεικτικά στοιχεία για το όλο ζήτημα της αηφορίας των καυσίμων, των βιοκαυσίμων. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Κομισιόν ουσιαστικά να συμβιβάσει τα συμφέροντα της βιομηχανίας, βιοκαυσίμων η οποία φυσικά έχει εύλογες προσδοκίες ε, Συμμετοχή ε, σε αυτή την επίτευξη του στόχου του 10% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το, η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι σήμερα γνωρίζουμε πω ε, κάποιες εκπομπές αφήνονται στο πλάι όταν εξετάζουμε τη μείωση αερίων θερμοκηπίου λόγω των βιοκαυσίμων και μερικέ φορέ ε, είναι σημαντικές ε, αυτές οι εκπομπές που παραγνωρίζονται και μερικές φορές και υψηλότερες από αυτές που υπολογίζουμε για τα ορυκτά καύσιμα. Τώρα τι κάνει η Κομισιόν, προσπαθεί να εξισορροπήσει αυτές τις δύο πτυχές. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι καλό θα ήταν να παγώσουμε την κατανάλωση συμβατικών βιοκαυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα επίπεδο ίσο με αυτό στο οποίο χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή η ανώτατη τιμή του 5%. Γι' αυτό συμπεριλάβουμε αυτό το 5% στην πρότασή μας. Είναι η σημερινή κατανάλωση εμπορικών βιοκαυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγγυόμαστε λοιπόν ότι οι παραγωγικές δυνατότητες που ήδη υπάρχουν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Ταυτόχρονα όμως σκεφτήκαμε ότι ο ορισμός ενός ανώτατου ποσοστού είναι ένα στιβαρό εργαλείο πολιτικής ε, για τον περιορισμό επιπλέον εκπομπών λόγω ε, έμεσης αλλαγής ε, χρήσης γης ε, εξαιτίας της χρήσης των σημερινών βιοκαυσίμων. Θεωρούμε ότι η επιστήμη ακόμα δεν βρίσκεται σε τέτοιο σημείο που να μπορεί να μας παράσχει την βεβαιότητα που χρειαζόμαστε για να συμπεριλάβουμε τους παράγοντες των βιοκαυσίμων στα κριτήρια αηφορίας όσον αφορά τις ζωοτροφές. Γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτό το ανώτατο όριο είναι ένα στιβαρό μέτρο σε σύγκριση με μια κατάσταση όπου θα χρειαζόταν να επανυπολογίζουμε διαρκώς τις εκπομπές με αποτέλεσμα ένα σταθές και αναξιόπιστο πλαίσιο για αυτές τις πολυπόθητες επενδύσεις στα βιοκαύσιμα. Επίσης ξεκινήσαμε θεωρώντας δεδομένο ότι ο Ευρώπης νομοθέτης δεν θα αγγίξει τους στόχους της οδηγίας ε, ποιότητας καυσίμων και ενέργειας. Η πρότασή μας λοιπόν βασίζεται κυρίως ε, στην ιδέα ότι παραμένει στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επίτευξη αυτών των στόχων και ότι γίνεται μια προσπάθεια κάλυψης του πιθανού κενού που θα δημιουργηθεί από αυτό το ανώτο του 5% παρέχοντας κίνητρα στα προηγουμένα βιοκαύσιμα. Αυτό θα διευκόλυνε τα κράτη-μέλη να επιτύχουν τους στόχους, διότι ένα κομμάτι της ενέργειας, μία μονάδα της ενέργειας από βιοκαύσιμα θα αντιστοιχεί σε δύο μονάδες προηγουμένων βιοκαυσίμων. Ε, αυτό θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να επιτύχουν το στόχο ακόμα και με το ανώτατο όριο. Η δεύτερη πτυχή αυτής της πολλαπλής μέτρησης θα ήταν ότι θα παρήχαμε πολύ συγκεκριμένα κίνητρα για την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση βιοκαυσίμων τα οποία παρουσιάζουν χαμηλό κίνδυνο εκπομπών. Ταυτόχρονα αυτό θα ενισχύσει την κοινοτομία και θα επιτρέψει σε όλες τις πολιτικές βιώσιμης, εν, ε, βιώσιμης ενέργειας μεταφορές να είναι πιο αξιόπιστες στη, στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών και θα συμβάλλουν στην ε, διαμόρφωση ενός σταθερού πολιτικού πλαισίου για τις αναγκαίες επενδύσεις ε, στο μέλλον, διότι τα βιοκαύσιμα θα μείνουν. Αυτό είναι σαφές όταν εξετάζουμε τον οδικό χάρτη για την ενέργεια εν ώψη του 2050 και μια οικονομία χαμηλής ε, ενέργειας. Χρειαζόμαστε βιοκαύσιμα, χρειαζόμαστε βιοκαύσιμα άλλα από αυτά που έχουμε σήμερα στην Ένωση, συνοπτικά η πρόταση της Επιτροπής θέτει το νέο μήνυμα που ούτως ώστε να περάσουμε προς τα προηγμένα βιοκαύσιμα και να μείνουμε αξιόπιστοι στους στόχους για, την, για τα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι κύριε Βίλς. vielen Dank.